so we, we, we, we vote. Yeah. Yeah. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, Dear colleagues, good morning. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε ε, τις εργασίες της Επιτροπής μας σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση στη συνάντηση των συντονιστών που προηγήθηκε και θα ανακοινώσω αργότερα τη σύνοψη των συζητήσεων των συντονιστών. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2011 κάθετος 11 ως προς την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα φορολογίας. Επομένως, παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας και να τις ε, βάλετε στη σχισμή, την ειδική. Καλώς. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 48 αποσύρθηκε. Καλώς. Θα ψηφίσουμε και τη 48, δεν είχα σωστές πληροφορίες. Ποιος είναι υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Απορρίπτεται. 'Δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 και 54 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά να το επιβεβαιώσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Κυρία Ντελβό, το δικό σας ε, λειτουργεί, δεν είναι η δική σας συσκευή. Καλώς. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε, ναι. Ας το ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 53, παρακαλώ. Απορρίπτεται. 11 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. εγκρίνεται. 11 προς 9, 11 υπέρ, 9 κατά. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές πρέπει να τα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 22 τροπολογία ψηφίζουμε. 10 προς 9 εγκρίνεται. 10 υπέρ 9 κατά. Δεν έχω τη κάρτα μου, αλλά είμαι υπέρ. Ψηφίζω υπέρ. Άρα 11 υπέρ 9 κατά. Καλώς. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. 23 με συγχωρείτε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Με συγχωρείτε εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε την 3. απορρίπτεται. 10 ε, κατά 9 υπέρ. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 37 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ Κατά. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 38 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Σαράντα. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, γιατί η 39 έχει διαγραφεί. Δεν θα, ψηφίσουμε τη 40 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται το σύνολο της νομοδότησης, στο σχέδιο. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του σχεδίου νομοδότησης. Συγγνώμη, πρέπει να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αυτό. Ψηφίζουμε επί του συνόλου. Εγκρίθηκε. 13 υπέρ 9 κατά μία αποχή. Συνεχίζουμε με την ψήφιση της έκθεσης Καρίμ. So, uh, compromise. Συμβιβαστική 1. Ψήφι πέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυκο 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αν 2 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 5 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 2 υπέρ κατά. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε την έμπλ 6 Επιτροπή Επασχόλησης, η 6. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται 8-12. 8, υπέρ 12 8 τροπολογία υπαριθμών 4, ψήφι υπέρ. Α, μισό λεπτό. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παραλείψαμε την τροπολογία 5. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, ψήφι υπέρ. Καταπίπτει. Ωραία. Ωραία. Συμβιβαστική 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επιτροπής Απασχόλησης 8 υπέρ και 19 τότε, υπέρ κατά. Κάποια σύγχυση βλέπω να έχει δημιουργηθεί. Ψηφίζουμε την ΑΦΚΟ 19. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 χωρίζεται σε δύο μέρη. Ψηφίζουμε υπέρ του πρώτου μέρους, κατά του πρώτου μέρους αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Για να κάνουμε έναν έλεγχο. Απορρίφθηκε. 11, 11, δύο αποχές. 11 ε, με συγχωρείτε, 2, 9 αποχές. Τι κάνουμε τώρα, ελέγχουμε, μετράμε 2 ψήφους του ΕΛΚ. Α, εντάξει. Εντάξει με την κάρτα. Ναι, ναι, είναι η πρώτη φορά που ψηφίζω με την κάρτα όμω. Ωραία, ωραία. Για να είμαστε σίγουροι επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 15. Δεύτερο μέρος της τροπολογίας 15. Ωραία. Εγκρίνεται. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε. Απορρίφθηκε. Κοντ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δώδεκα. Έμπλ υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 14 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάει στη συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά σκάνουμε έναν έλεγχο απορρίφθηκε Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση Απορρίφθηκε. Τροπολογία 34. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίφθηκε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελέγχουμε το 35. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές να απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αύκο 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. αυκο 7. αυκο 10 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται αυκο 12 υπέρ κατά για να κάνουμε έναν έλεγχο Εγκρίνεται. Αμπλένα. Εμπλένα. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εμπλ 4. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εμπλ 10. Υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. Κοντ 2. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Κον 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. κοντ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. κοντ 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. κοντ 9 υπέρ. Κατά για να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Κοντ 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, κοντ 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τα δύο υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση Είναι τα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Για μισό λεπτό. Για να βεβαιωθούμε. Ένας ακόμα. Ένας ακόμα. Ωραία. Εγκρίνεται, εγκρίθηκε. Είναι τα τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την... Ε, είναι τα 4 είναι τα Εγκρίθηκε. Ωραία, εγκρίθηκε. Είναι τα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και έκθεση στο σύνολό του. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Για να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Εγκρίθηκε λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε Καρένη. Uh, now, we have Mrs. If Mrs. McGuinness is, she is here. We, yes. we have uh, Mrs. McGuinness here. Η κυρία Μαγκρίς είναι εδώ. Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω το, το λόγο σχετικά με το θέμα που συζητήθηκε χθε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την κατανόηση που δείξατε αφήνοντάς με να μιλήσω σήμερα στην Επιτροπή μετά από τη χθεσινή ακρόαση. Η νύχτα υπήρξε καλός σύμβουλος και ελπίζω ότι θα βοηθήσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ που λάβατε αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν σημαντικό να οργανώσει η Επιτροπή την ακρόαση χθε. Ο ρόλος μου ως Ευρωπαίου ε, διαμεσολαβητή σε θέματα απαγωγής παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικός και στόχος είναι να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι εφαρμόσιμη για την οικογένεια, πάντοτε έχοντας κατά νου τα συμφέροντα του παιδιού. Συνεπώς το θέμα το βλέπω από αυτή την οπτική γωνία. Όπως ε, γνωρίζετε, το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο. Ο αριθμός των μεικτών γάμων αυξάνεται και ξέρουμε ότι 200 250.000 παιδιά αναφέρονται ως αγνοούμενα κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 36% είναι θύματα απαγωγής. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε γενικές γραμμές, αν κοιτάξουμε το θέμα στα πλαίσια του κανονισμού Βρυξέλλες 2, οδηγούμεθα στο να ξεπεράσουμε μερικά από τα προβλήματα της Σύμβασης της Χάγης και ως ένα βαθμό τα καταφέρνουμε. Θα ήθελα όμως εν συντομία να αναφερθώ στην, σε συγκεκριμένη εμπειρία. Έχουμε ένα δείγμα 90 περιπτώσεων που εξετάσαμε στους τελευταίους 12 μήνες. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες πτυχές που αφορούν πρακτικά και νομικά προβλήματα. Για παράδειγμα, μερικά από τα νομικά θέματα. Σύγκρουση των ε, νομολογιών, θέματα επιμέλειας του παιδιού, ε, θέματα τα προβλήματα ορισμού σε ό,τι αφορά τη συνήθεια κατοικία, παραβίαση του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη, ακρόαση, επιπλοκή εκεί που οφείλονται ε, σε, οφείλονται σε καθυστερήσεις. Μερικά από τα πρακτικά θέματα που τίθεται αφορούν διοικητικέ καθυστερήσεις σε επίπεδο αστυνομία ή ε, ε, σε επίπεδο δικαστικό, προβλήματα στην εφαρμογή των δικαιωμάτων επικοινωνίας με το παιδί, προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των γονιών και του παιδιού. Αν τώρα κοιτάξουμε τον κανονισμό, το θέμα που ανακύπτει διαρκώς αφορά συγκρούσεις σχετικά με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και προβλήματα εφαρμογής από το δικαστήριο μιας άλλης χώρας μέλου. Υπάρχει το θέμα βεβαίως της συνήθους κατοικίας. Για παράδειγμα, στην, τον κανονισμό Βρυξέλλες 2, ο όρος συνήθης κατοικία δεν ορίζεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ κάποιο τηλέφωνο χτυπάει, λέει η κυρία πέστε τους ότι δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ωραία. Το δικαστήριο συνεπώς συνεχίζει να είναι αρμόδιο μέχρι τη στιγμή που το παιδί θα εγκατασταθεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε όμως περιπτώσεις όπου έχουν δικαιοδοσία και τα δύο δικαστήρια λόγω του ασαφούς προσδιορισμού του όρου συνήθις τόπος κατοικίας. Και βεβαίως ε, ε, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και συγκρούσεις. Και για ένα παιδί η καθυστέρηση είναι μείζον πρόβλημα. Αν λοιπόν θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο παιδί, θα πρέπει να κατανοήσουμε την επίπτωση που έχει αυτό στο παιδί ή στα παιδιά. Πραγματικά πιστεύω ότι το θέμα της συνήθους κατοικίας, συνήθους τόπου κατοικίας θα πρέπει να ρυθμιστεί και θα πρέπει να υπάρχει άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως και η δική μας εμπειρία είναι ότι η απόφαση ενός δικαστηρίου δεν εφαρμόζεται άμεσα ή σωστά σε μια άλλη χώρα. Ε, έγινε μια μελέτη σχετικά με την ε, δικαστική επαγωγή παιδιών και μας δείχνει ότι η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων ε, μιας χώρας θα πρέπει να ξεκινάει από τις πρώτες φάσεις και μερικές φορές η άμεση επαφή μεταξύ των δικαστών θα μπορούσε να συμβάλλει στο να ξεπεραστούν μερικά προβλήματα που οδηγούν σε καθυστερήσεις στις ε, ε, αποφάσεις. Και αυτό έχει άμεση επίπτωση στα παιδιά. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω στο θέμα της διαμεσολάβησης γιατί και πάλι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό θέμα. Πριν αναφέρω τόσο ορισμένα θέματα που αφορούν τη διαμεσολάβηση, θα ήθελα περιληπτικά να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που επιδέχονται βελτιώσει. Για παράδειγμα, ε, το πλαίσιο για την υποβολή ε, εντάσεων. Εκεί χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών. Αυτό είναι ένα θέμα ε, που θα μας απασχολήσει. Σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση, κατάλαβα ότι απασχολούν σπένες τεχνικές και νομικές πτυχές του κανονισμού, γιατί στόχο έχουν να διαφυλάξουν τα παιδιά και την, ε, να μην διονύσουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Το θέμα λοιπόν της διαμεσολάβησης ε, θα μπορούσε να ε, έχει πολλά ωφέλη για όλα τα μέρη. Βεβαίω δεν είναι μια μαγική φόρμουλα, αλλά ε, είναι ένας ε, τρόπος ε, για τους γονείς να βρουν μια λύση για τις οικογένειές και τα παιδιά τους αντί να επιβάλλει μια λύση στην κατάσταση το δικαστήριο. Συνεπώς οι συμφωνίες και, των, και από και των δύο γονιών είναι πιθανότερο να καταλήξουν σε ένα καλό αποτέλεσμα μακροχρόνια. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Βεβαίως η μελέτη που έγινε το 2012 σχετικά με τις απαγωγές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν την ενδυνάμωση των μέτρων που αφορούν τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις απαγωγής παιδιών. Ιδιαίτερα η μελέτη Apple λέει ότι θα πρέπει να γίνουν τροπολογίες, τροποποίηση των κανονισμών και να συστηθούν ζητούν προληπτικά προγράμματα διαμεσολάβησης. Αυτό μετά σαν αποτέλεσμα της οδηγίας που ψήθηκε το 2004 και που αφορά το ρόλο του διαμεσολαβική όταν έχουμε να κάνουμε με ε, παιδιά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα της διαμεσολάβησης σε αυτό το πλαίσιο. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο για να ενθαρρύνουμε τα δικαστήρια να στραφούν προς την διαμεσολάβηση μεταξύ των ε, μερών. Ε, θα πρέπει ε, λοιπόν να ενδυναμωθεί ο ρόλος της διαμεσολάβησης γιατί ενδεχομένως οδηγεί σε μία μεγαλύτερη δέσμευση. Ενδεχομένως το θέμα αυτό είναι υποσυζήτηση, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει συμφωνία σχετικά με το ρόλο της διαμεσολάβησης και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει στην αθεώρηση του κανονισμού. Ξέρω ότι χθε η Επιτροπή μίλησε για την, ε, το να αποκτήσουν ένα κεντρικό χαρακτήρα τα δικαστήρια που ασχολούνται με περιπτώσεις απαγωγής παιδιών. Αυτό είναι βέβαια κάτι σαφώς καλοδεχούμενο γιατί τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα αλλά θα μπει και ένα χρονικό πλαίσιο. Οι δικαστές και όχι οι δικηγόροι που συνεργάζονται στενά με τους διαμεσολαβητές είναι ένα θέμα που επίση θα πρέπει να μα απασχολήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το ρόλο που παίζουν οι διαμεσολαβητές και το ρόλο που παίζουν αυτοί που κινούνται σε επίπεδο νομικό. Και βεβαίω και για τους δύο απαιτείται κατάρτιση. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά ενδυναμώνοντας τα μέτρα που προβλέπει ο κανονισμό, καταρτίζοντας περαιτέρω τους δικαστές και τους διαμεσολαβητές και συνεργαζόμενοι με συνεργασία με τις κεντρικές αρχές ε, και τους αντιμεσολαβητές. Βεβαίως όλοι ε, έχουμε κατά νου το συμφέρον των παιδιών και ο κανονισμός των Βρυξελών μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να βελτιώσουμε τα πράγματα στους τομείς αυτούς που ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως παραμένει η πολυπλοκότητα του ε, νομικού συστήματος αλλά παρόλα αυτά στο παιδί και στην οικογένεια θα πρέπει να δώσουμε ό,τι καλύτερο σε θέματα επιμέλειας και θα πρέπει να πω ότι η διαμεσολάβηση θα μπορέσει να έχει κάποιο αποτέλεσμα εάν, συμβεί, εάν λάβει χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο. Για παράδειγμα, εγώ ασχολήθηκα με δύο περιπτώσει διαμεσολάβηση του τελευταίου δύο μήνε. Σε ορισμένε περιπτώσει δεν τα καταφέρνουμε καθόλου, γιατί φτάνουν στα χέρια μα πάρα πολύ αργά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Αλλά όταν τα μέρη είναι διατεθειμένα να συζητήσουν, θα μπορούσε αυτό να αποβεί προ όφελο όλων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, madam, for your... Σας ευχαριστώ πολύ, για τις συμβατικές υποδείξεις σας σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Εσείς μέλη έχετε ερωτήσεις? Κανείς δεν έχει ερώτηση. Ευχαριστώ λοιπόν που μοιραστήκατε τις απόψεις σας μαζί μας. Ο πρόεδρος συνεχίζει. Θα προχωρήσουμε στο υπαριθμό 11 και την κυρία Ντελβό για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και επιχειρήσεων με την απλοποίηση ορισμένων δημοσίων εγγράφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ίσως ότι βρισκόμαστε σε τριμερή διάλογο. Ήδη σήμερα το απόγευμα προβλέπεται τριμερή διάλογος και ίσως μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Τα ζητήματα που είναι σημαντικά για το Κοινοβούλιο, δηλαδή, τα υπενθυμίζω, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απέχει πολύ από την θέση του Συμβουλίου διότι μιλούμε για κατάργηση της επισημείωσης και της νομιμοποίησης και σε πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο είχε περιλάβει μεγάλο αριθμό εγγράφων στο πεδίο εφαρμογή. Το Συμβούλιο ε, με τη σειρά του μετά από μακρές συζητήσεις που διαρκούν ήδη μια τετραετία συμφώνησε επί μια σύντομη λίστας δημοσίων εγγράφων που αναφέρονται μόνο στα προσωπικά δεδομένα, γέννηση, θάνατο, γάμο ή εταιρική σχέση. Συζητήσαμε δε διαμακρών με το Συμβούλιο. Επιμικίναμε πάλι τον κατάλογο, προσθέσαμε δηλαδή τρία δημόσια εγγραφά στον κατάλογο. πιστοποιητικό βίου, ένα έγγραφο που επιτρέπει σε ένα πολίτη να πάει να ψηφίσει σε άλλη χώρα από αυτήν της οποίας έχει την ηθαγένεια και τρίτο η... το ποινικό μητρό. Επίσης μπορέσαμε να επιμικίνουμε την λίστα των πολυγλώσσων εγγράφων. Στην αρχή το Συμβούλιο είχε προτείνει μόναχα τέσσερα. Τώρα έχουμε φτάσει σε δέκα περίπου πολύγλωσσα έγγραφα τα οποία θα συναπαρτίζουν μέρος του εγγράφου. Προσπαθήσαμε να περιλάβουμε ακόμα περισσότερα εγγραφά στο πεδίο εφαρμογή και τελικώ συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο ένα είδο επανεξετάσεω. Δύο χρόνια δηλαδή μετά από τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια μελέτη επιπτώσεων έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ενδεχομένως στο πεδίο εφαρμογής τα έγγραφα που αναφέρονται στις επιχειρήσεις, δηλαδή στο καθεστώς μιας επιχειρήσεως και το καθεστώς του εκπροσώπου της επιχειρήσεως, καθώς και έγγραφο για τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και πανεπιστημιακά ε, πτυχία κλπ. Καθώς επίσης και για την πιστοποίηση αναπηρίας, που και αυτό δεν θα χρειάζεται πλέον επισημείωση. Έχουμε δύο θέματα τώρα ακόμη, αφενός την υποχρέωση ενημερώσεως, θέλουμε να περιληφθεί μια ξεκάθαρη υποχρέωση των χωρών μελών να πληροφορούν τους πολίτες, ότι δηλαδή ο πολίτης εφόσον έρχεται να ζητήσει επισημείωση ότι δεν απαιτείται επισημείωση εφόσον το έγγραφο απευθύνεται σε άλλη χώρα μέλος της Ένωσης. Και δεύτερον, σχετικά με τα έξοδα. Ιδίω τα ε, πολύγλωσσα έγγραφα ποια είναι τα έξοδα για την ε, ε, κτήση των εγγράφων αυτών. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε κοντά πια σε μια συμφωνία, θα δούμε βέβαια το απόγευμα. Ένα πράγμα με εξέπληξε στις ε, συζητήσεις, αφενός η μεγάλη δυσπιστία μεταξύ τους. Δηλαδή καμία χώρα δεν εμπιστεύεται τα δημόσια έγγραφα της άλλης χώρας. Βεβαίω έτσι αυτό το θέμα γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Παρόλο που η επίθεση επισημειώσεως από το Υπουργείο Εξωτερικών σε ένα έγγραφο του δίνει βέβαια κάπως επίσημο χαρακτήρα, αλλά δεν αποδεικνύει τίποτε, ενώ με το νέο σύστημα που προτείνουμε, το ΙΜΙ δηλαδή, εφόσον η δημόσια διοίκηση μιας χώρας μέλους έχει αμφιβολίες για την γνησιότητα του επισήμου εγγράφου, το βάζει στο σύστημα και αμέσως έχει απάντηση από την ε, ε, αρχή του άλλου κράτου εάν το έγγραφο που έχει εκδώσει είναι πράγματι γνήσιο ή Έτσι λοιπόν θα ενισχυθεί το σύστημα. Άρα βέβαια ε, ανατρέπει κάποιες συνήθειε. Αυτά λοιπόν οφείλονται σε μια στάση του Συμβουλίου που λέει μα έχουμε τη συνθήκη της Χάγης. Είναι ανάγκη τώρα να φτιάξουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία που μάλιστα θα αντίκειται στην ε, συνθήκη της Χάγης ή Σύμβαση Δεν υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενθουσιασμό από πλευρά Συμβουλίου Υπουργών να εφαρμόσουν το, το, τη ρύθμιση αυτή και γι' αυτό νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια η οποία έχει προτείνει ένα κείμενο εμείς σκεπτόμαστε τους πολίτες αν θέλουμε πραγματική ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και των εμπορευμάτων, διότι μιλούμε βεβαίως για ενιαία αγορά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να καταργήσουμε όλες τις περιτές τυπικότητες, ε, τυπικές διαδικασίες που ως είναι περιτές επαναλαμβάνω. Ελπίζω όπως είπα ότι θα καταλήξουμε σε συμβασμό σήμερα το απόγευμα. Ιδού λοιπόν αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια από τα μέλη. Δεν βλέπω κανείς να ζητάει το λόγο. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντελβό. Προχωρούμε με το σημείο 13. Εξέταση των ε, τροπολογιών της έκθεσης προς μια ενιαία ψηφιακή αγορά και αν κατάλαβα καλά ο εισηγητής κύριος Τζαμπάσκι ε, αντικαθίσταται από τον κύριο Λιούαρ. Έτσι δεν είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι συντονιστής από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Με λένε Άντριου Λιούερ και ασχολούμαι με την έκθεση αυτή. Ο κύριος Τζαμπάσκη μου ζήτησε εν συντομία να τον εκπροσωπήσω εδώ. Ζητά συγγνώμη διότι δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί σας και ε, δεν θέλει να μετατεθεί για άλλη ημέρα η συνεδρίαση. Και τα βασικά σχόλια ε, έχουν ως εξής. Κάθε φορά που θα λέω εγώ σε πρώτο πρόσωπο εννοώ ο κύριος Τζαμπάσκι. Λέει λοιπόν ο κ. Τζαμπάσκη τα εξή. Χαίρομαι διότι τόσοι πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και υπέβαλαν τροπολογίε, κάτι το οποίο θα ενισχύσει την ε, συμβολή τη Επιτροπή μα στην έκθεση ίδια πρωτοβουλία τη ΙΜΚΟ και τη ΙΤΡΑ. ΙΤΡΕ, συνεχίζω να αναλύω τι ε, τροπολογίε και στο Στρασβούργο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τι συμπληρωματικέ τροπολογίε εν ώψη τη πληροφορία του Νοεμβρίου λόγω του ότι υπάρχουν περιορισμοί στο, στις λέξεις στο ανώτατο χρονικό, στο ανώτατο όριο λέξεων και στη διατύπωση, θα προσπαθήσω να πετύχω τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Και κάθε τροποποίηση του πλαισίου για το copyright θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη και να ε, βοηθά στην ε, ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, να ενισχύει την εμπειρία του καταναλωτή, να βελτιωθούν οι διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, να υπάρχει streamlining, ευθυγράμμιση και ψηφιοποίηση των ε, απαιτούμενων για τις επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μικρόφωνο του ομιλητή, α, ευχαριστούμε, συγγνώμη, ε, ναι, το ίδιο ισχύει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το διασυνοριακό εμπόριο και τις αθέμητες τιμολογιακές διαφορές στο διαδίκτυο με βάση την εγκατάσταση, το που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, αλλά και ε, η οδηγία για τις υπηρεσίες. Όλα αυτά ε, πρέπει να συμβάλλουν προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι και η, η κατάλληλη ανταμοιβή για τους δημιουργούς περιεχομένου. Έχουμε τη συνθήκη ή τη σύμβαση του Μαρακές, οι συναδελφοί τη στηρίζουν ε, με σκοπό να στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρίες. Εξαιρέσεις, περιορισμοί θα πρέπει να είναι ε, ισορροπημένες και θα πρέπει πάντοτε να συμβάλλουν στη διευκόλυνση της καινοτομίας. Τα τέλη πνευματικής ιδιοκτησίας, copyright, από τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι ε, δίκαια και Έχουμε τους παρόχους διαδικτύου, υπηρεσιών διαδικτύου και τους μεσολαβητές, τους ενδιάμεσους και θα πρέπει οπωσδήποτε να εμπλακούν στη συζήτηση. Το ενοχικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Με στόχο να τονίσουμε ότι το δίκαιο αυτό πρέπει να συνάδει με την υφιστάμενη νομοθεσία, να αναγνωρίσει τις διαφορές μεταξύ ψηφιακού περιεχομένου και άλλου είδους περιεχομένου. Ε, δίκαιο συμβάσεων λοιπόν στο ψηφιακό κόσμο και ε, περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Έχουν ομαδοποιήσει οι σκιώδεις εισηγητές τις τροπολογίες τους, ε, κυρίως ως προς το πλαίσιο, το γενικό πλαίσιο για το copyright, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αντιγραφής και πιο συγκεκριμένες προτάσεις επίσης για προσβασιμότητα και φορητότητα διασυνοριακή. Ως προς το copyright, εξαιρέσεις προβλέπονται στις τροπολογίες που ζητούν εναρμόνιση των τελών copyright συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής αντιγραφής και του αντικτύπου που θα έχει αυτό στους ε, καταναλωτές. Το ISP, οι Internet Service Providers, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και η ενδιάμεση ε, θα πρέπει να ορίζονται σαφέστατα τα καθήκοντά τους, να υπάρχει ορισμός ε, του τι εστί ενδιάμεσος ή διαμεσολαβητής, τι για να υπάρχει σωστή κατανομή των ευθυνών. Δεν θέλουμε να προλάβουμε εξελίξεις τις οποίες επιζητά ε, επιζητούν οι καταναλωτές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε μία αναλογική προσέγγιση ε, στις ε, τροπολογίες που υποβάλλουμε και να γνωρίζουμε, να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση Διάφορες τροπολογίες ασχολούνται με την επιβολή του copyright, το εμπορικό σκέλος, τη συνειδητοποίηση, την λογική προσέγγιση, το ρόλο του παρατηρητηρίου. Να έχουμε υπόψη μας ότι ε, πρέπει στο copyright να μην μπαίνουν μόνο οι υπηρεσίες, αλλά να μπαίνουν και τα αγαθά, για να μην υπάρχουν παραθυράκια στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Τώρα, ως προς το ε, δίκαιο για τις συμβάσεις, Έχουμε διάφορες επιλογές και θα δούμε τους χειώδεις εισηγητές αν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμό, συμβαστικές τροπολογίες. Άλλες, κάποιες τροπολογίες θέλουν την πλήρη έγκριση, άλλες θέλουν ε, σημείο κίνησης να είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά την πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, λέει ο κ. Τζαμπάσκη, ε, για το ενδιαφέρον τους για την νομοδότηση αυτή και ανυπομονεί ο κ. Τζαμπάσκι να ε, συνεργαστεί με όλους εσάς έτσι ώστε η δική μας Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να συμβάλλει αποφασιστικά στη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ η κυρία Ρέκνερ. Ευχαριστώ τον εισηγητή Κέριγκερμαν. Εκτιμώ ιδιαίτερο, κυρία Ρέντα, με συγχωρείτε. Εκτιμώ ιδιαίτερο ε, όλα αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα μιας επιτροπής ε, για θέματα τα οποία είναι πολύ πολυσχηδή Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για το θέμα αυτό και είναι καλό που καλεί τη δική μας Επιτροπή να συμβάλλει στη συζήτηση. Υπάρχουν θέματα λογισμικού, υπάρχουν θέματα πληροφόρησης, υπάρχουν θέματα copyright και μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και αυτό είναι καλό. για το, την κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να πάρουν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούγοντας τον εισηγητή βλέπω ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες ωστόσο μακρόν έχουμε συζητήσει. Πράγματι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις και στη φορητότητα και στη διασυνοριακή πρόσβαση. Πώς όμως θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αυτή την φορητότητα, αυτό θα σημαίνει σημαίνει ότι το άτομο μεταφέρεται και μετακινείται και ταξιδεύει μέσα στη δική του νομική φούσκα κλεισμένος, δηλαδή ε, μεταφέρει τα νομικά δικαιώματα του κράτους στο οποίο υπάγεται όπου και να πάει. Αν πρόκειται να έχουμε φορητότητα, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα πρέπει να ε, αναγνωρίζεται να υπάρχει ταυτοποίηση του καθενός με πολύ προσωπικά στοιχεία και προσωπικές πληροφορίες και εκεί υπάρχει σύγκρουση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εάν πρόκειται να βελτιώσουμε τη διασυνοριακή πρόσβαση, τότε ποιο νομικό μέσο είναι το καλύτερο να χρησιμοποιηθεί. Έχω το βάλει τροπολογίες λοιπόν όπου έχω προτάσεις να δούμε ε, επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση μεταξύ άλλων, έτσι ώστε να περιλάβει το online demand, το video on demand και διάφορες άλλες ψηφιακές υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας. Και ξέρουμε και ποιες εξαιρέσεις και ποιοι περιορισμοί τώρα είναι οι πιο κατάλληλοι να δούμε τι συζητήσεις είχαμε και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, Πολλοί συζητήσαμε το διαχωρισμό ε, της εμπορικής από τη μη εμπορική χρήση στη συζήτηση για την ελευθερία του πανοράματος και είδαμε ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πολύ λειτουργικό στην πράξη γιατί δεν συνάδει ούτε με τις προσδοκίες ε, των χρηστών για το τι εστί εμπορικό και το τι δεν εστί εμπορικό. Λοιπόν, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη και να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για αυτό το οποίο θέλουμε να επιτρέψουμε. Δεν νομίζω ότι οι μη εμπορικοί περιορισμοί είναι ε, χρήσιμος τρόπος να πετύχουμε το στόχο μας. Άλλωστε έχουμε ήδη προβλήματα με αυτό του είδους το διαχωρισμό. Αλλά και στο θέμα της επιβολής της νομοθεσίας δεν υπάρχει λόγος να επανεφεύρουμε τον τροχό το Κοινοβούλιο έχει ήδη καλωσορίσει την προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της και θα πρέπει να δώσουμε χρόνο να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο δράση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι ανάγκη να έχουμε περισσότερα στοιχεία στο θέμα των δικαιωμάτων αντιγραφή copyright και άλλων δικαιωμάτων διανοητική ή πνευματικής ιδιοκτησίας και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο έτσι ώστε να υπάρξουν τέτοιου είδου αποδεικτικά και άλλα στοιχεία. Θα ήθελα να τονίσω ε, και την τροπολογία για την προειδοποίηση notice and takedown. down. Διαδικασίες δηλαδή προειδοποίησης ενημέρωσης και ε, ε, αφαίρεσης από το διαδίκτυο του εκάστοτε περιεχομένου. Πώς θα δουλέψουν όλα αυτά εάν δεν έχουμε εναρμόνιση των δικαιωμάτων αντιγραφής copyright. Εάν για παράδειγμα μια εταιρεία πρέπει να αφαιρέσει μία ιστοσελίδα γιατί ε, της έχει κοινοποιηθεί ότι υπάρχει παράβαση. Ε, ποια εξαίρεση copyright θα εφαρμόσει αυτή της δικής της χώρας ή την εξαίρεση copyright ε, της χώρας από την οποία ήρθε η γνωστοποίηση και η ειδοποίηση. Σε τέτοιου είδους λοιπόν διαδικασίες, notice and take down, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ακυρώνονται γιατί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, δεν είναι οι ίδιοι στην Ευρώπη και δεν ε, ε, είναι σαφές ε, ποιοι πρέπει να εφαρμοστούν, ποιας χώρας δηλαδή. Από τη μία υπάρχει μια ευρεία ε, διασυνοριακή διάσταση και εκεί θα πρέπει να έχουμε εναρμόνιση όσο το περισσότερο. Από την άλλη υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι ε, φορείς ε, λειτουργίας, εκμετάλλευσης, intermediaries. Πράγματι χρειαζόμαστε ένα νέο ορισμό όλων αυτών. Και αυτός ο νέος ορισμός υποκρύπτει και πολλούς κινδύνους αν θέλετε γιατί ο ε, ορισμός που έχουμε σήμερα έχει λειτουργήσει αρκετά καλά με βάση την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να δούμε και τις διαβουλεύσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ευθύνες ε, των ενδιάμεσων φορέων και να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη στη διάθεσή μας. Τέλος, για τα τέλη. Αυτό είναι και ο μεγάλος ελέφαντας μέσα στην αίθουσα για τον οποίο δεν μιλάει κανείς τα θέματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς διότι από τη μία είναι εξαιρετικά δύσκολο να εναρμονιστούν τα τέλη γιατί το κάθε κράτος μέλος έχει δική του προσέγγιση από την άλλη όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ότι υπάρχουν διαφορετικά τέλη ή φόροι ε, στα προϊόντα στις διαφορετικές χώρες είναι και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ενιαία ψηφιακή αγορά και θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε όλο και περισσότερη εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Δεν αποτελεί εξαίρεση π.χ. Αντιθέτως, συνήθι πρακτική αποτελεί το γεγονός οι κατασκευαστές προϊόντων να πρέπει να πληρώσουν τέλη και φόρους για το ίδιο προϊόν δύο φορές όταν αυτό ταξιδεύει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τελικά ποια, ε, ποιος είναι ο αρνητικός αντίκτυπος από το private copy, από την ιδιωτική αντιγραφή, εάν υπάρχει, και να φτάσουμε σε μια κατάσταση κατά την οποία ο υπολογισμός της ζημίας, της βλάβης, ε, γίνεται με σταθερά, με στέρεα στοιχεία. Αυτά προς το παρόν είναι τα σχόλιά μου. Προσδοκώ με ανυπομονησία να συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους λοιπούς σκιώδεις εισηγητέ. Νομίζω ότι πράγματι η Επιτροπή μας μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά, να ε, έχει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο απτές και συγκεκριμένες κατευθύνσεις και υποδείξεις για το πώς θα εφαρμόσει ε, τα μέτρα στους ε, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και λοιπούς σε θέματα copyright και άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Λούερ για την έκθεση αυτή η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπω με χαρά ότι το θέμα των απολαμβών των δημιουργών αναφέρεται στην έκθεση γιατί αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχουμε τα δικαιώματα αντιγραφής, το copyright γιατί δίχως αυτό δεν θα υπήρχε καμία προστασία για τους δημιουργούς. Και αν δεν υπάρχει προστασία, γιατί ποιο λόγο το κάνουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια αναφορά στην συνθήκη του Μαρακέσα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς. Όταν συζητήσαμε και ψηφίσαμε την έκθεση της κυρίας Ρέινταρα, ασχοληθήκαμε πολύ με το όλο θέμα των περιορισμών και των εξαιρέσεων που συμφωνώ είναι ένα δύσκολο θέμα Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω σε ό,τι αφορά το θέμα της εναρμόνισης των εξαιρέσεων και των περιορισμών. Γιατί ο νόμος για το copyright και τα συστήματα στις διάφορες χώρες μέλη διαφέρουν. Και νομίζω ότι το να αναμένουμε πλήρη εναρμόνιση δεν είναι κάτι εφικτό. Αυτό που κατέστησε σαφέ στην έκθεση Radar, κάτι που συμφώνησε και το Κοινοβούλιο, είναι το θέμα των ελάχιστων προτύπων. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν σε ορισμένου τομεί εναρμόνιση και περιμένουμε να το κάνει και κάθε χώρα μέλο. Πράγματι, οι τομεί αυτοί είναι η, εξαίρεση, η εκπαίδευση που είναι μια εξαίρεση στι περισσότερε χώρε. Αυτό είναι πρακτικό, μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η κυρία Ρέινταρα, νομίζω τα ελάχιστα πρότυπα είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και ακριβώς έτσι θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω το όλο θέμα, δηλαδή οι διακρίσει σε επίπεδο εμπορικό, είναι δύσκολες και μιλάμε για νέους ε, ε τομείς. Ας πούμε ενέβρεση δεδομένων, ε, αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο και θα υπάρξουν όλο και περισσότερα σε αυτό το τομέα με την βελτίωση της τεχνολογίας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να θέσουμε ορισμένα ελάχιστα πρότυπα. Υπάρχουν ε, δυσκολίες, μία από τις δυσκολίες της ψηφιακής αγοράς είναι ότι κινείται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Συνεπώς χρειαζόμαστε κάποιον τρόπο για να μπορούμε να αποδείξουμε ορισμένα πράγματα για να, για να μπορέσουμε να έχουμε ορισμένες νομικές βεβαιότητες. Διαφορετικά δεν θα είναι τα πράγματα, δεν θα τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε στην έκθεση Radar. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για, και για ορισμένε ενδιάμεσε πλατφόρμες. Ξέρω ότι η Επιτροπή έχει σκοπό να υποβάλει μία πρόταση σχετικά με αυτό το θέμα. Πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι οι ενδιάμεσοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Θα πρέπει πραγματικά να έχουμε τη βεβαιότητα ότι κινείται καλά η αγορά αυτή, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μερικοί από αυτούς ε, δεν συμφωνούν τόσο πολύ και με τους κανόνες και τους κανονισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι μία από τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι οι ανταμείβονται όπως θα έπρεπε και θα πρέπει να υπάρξουν και ελάχιστα πρότυπα. Αυτό είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριος Μάουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί πολλά από τα θέματα θίγησαν ήδη από τους συναδέλφους. Εγώ πρότεινα μία σειρά από τροπολογίες που κατ' ουσία προβάλλουν ορισμένες ιδέες για την εναρμόνιση του συστήματος copyright, ας πούμε το σύστημα της ε, ε online. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να διακυβευτεί η τοπική ταυτότητα. Θα ήθελα επίσης να προτείνω ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα μεγαλύτερης συνεργασίας με όλους όσους έχουν σχέση με αυτό τον κλάδο. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο νομικό περιεχόμενο που αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλο το δίκτυο. Και θα πρότεινα να γίνει και μία αναθεώρηση του ενδιάμεσου online έτσι ώστε να μπορέσει να διευκρινιστεί η ευθύνη του που θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά τα ε, συγγραφικά δικαιώματα και το πώς θα μπορούν να ορίζονται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων με αποτελεσματικότητα. Αυτά. Αυτό είναι το, η, βασική, ουσία των τροπολογιών που υπέβαλα. Ευχαριστώ κύριο Σιέφκα. Ε, ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία-δύο παρατηρήσεις εξ ονόματος του σκιώδου συζητητή του κυρίου Ράντεπ που σήμερα δεν τα κατάφερε να είναι εδώ. Το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεών του ευθυγραμμίζεται με αυτά που είπε ο εισηγητής γνωρίζω, ότι ο εισηγητής επικοινωνεί και με τους άλλους ε, σχεδόν εισηγητές. Εδώ μιλάμε όλοι για το δυναμικό της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και νιώθουμε την ενέργεια που έχει αυτό. Το θέμα είναι τα μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε καλά αυτό το δυναμικό Σκέφτομαι ιδιαίτερα αυτούς τους οποίους απευθύνεται αυτό το δυναμικό, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους επιχειρηματίες που δίχως άλλο αναμένουν ένα και μοναδικό πράγμα από μας, το να έχουμε ένα διαφανές, να τους ε, παραδώσουμε ε, ένα μέσο διαφανές που θα περιγράφει με σαφήνεια τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Συμφωνώ με τον κύριο Χάνιβαλ. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά διαρκώς εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί κανείς ε, να την παρακολουθήσει. Μερικές ε, φορές οι οδηγίες δεν είναι τόσο ε, λεπτομερής. Πέρα όμως από τα θέματα της διαφάνειας, εμείς ε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε αυτές οι διατάξεις να είναι σωστές για όλους τους χρήστες και για τους διανομής, τους παραγωγούς, για τους καταναλωτές, για τους χρήστες, για όλους τους φορείς εκείνους που εμπλέκονται σε αυτές τις δράσεις. Βεβαίως έχουμε απόλυτη συνείδηση του ότι στα πλαίσια Τη στρατηγική που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μα Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος του νομοθετικού πακέτου. Από εμά θα εξαρτηθεί ε, το κατά πόσον θα υπάρξει αυτή η μετακίνηση. προς μία πιο αποτελεσματική χρήση της ιδιακής αγοράς της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν ε, να θέσουμε ορισμένα θέματα. Μερικά από αυτά έχουν ήδη τεθεί. Θα είναι αναγκαία η φορητότητα ε, ε, του περιεχομένου. Είναι σημαντικό αυτό γιατί αυτή η φορητότητα θα δημιουργήσει σύγκληση μεταξύ των χρηστών, μεταξύ των καταναλωτών και του το κλάδου, του τομέα της δημιουργίας. Από την άλλη πλευρά θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ορισμένα νομικά θέματα διαδικτυακά. Αυτό είναι κάτι που περιμένουν όλοι και θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο, σαν ε, όπως θεωρούμε δεδομένο το ότι αναπνέουμε. Η αποτελεσματική χρήση όλων αυτών των μέσων συνδέεται και με τα συγγραφικά δικαιώματα, με το copyright που είναι πολύ λογικό. Ελπίζουμε κάποια στιγμή θα αποτελέσει τη βάση για κάθε δημιουργική δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να προσανατολιστεί, να έχει στόχο την βελτίωση της λειτουργίας, επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε ε, για την προστασία των δικαιωμάτων. Αυτό κατά τη διάρκεια όλης της αλυσίδας, κατά μήκο όλης της αλυσίδας που συνδέει το δημιουργό με τον διανομέα και τελικά με τον καταναλωτή. Αυτό θα βοηθήσει στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Εγώ συμφωνώ με όσα υπόθηκαν ως προς την ανάγκη της προστασίας των πολιτιστικών διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μέσα από την χρήση της αρχής της εδαφικότητας μια αρχή που προστατεύει την πολιτιστική διαφορά στα πλαίσια των εργασιών που έχουμε να κάνουμε. Μιλώντας για το δικαίωμα αγοραπολισίας, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το μέσο. Αυτό είναι το νομικό μέσο που έχει το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς μεταξύ των οποίων και της ψηφιακής αγοράς. Η αύξηση των διαδικτυακών πολίσεων είναι δυνατή μόνον αν έχουμε σαφείς διατάξεις. Αυτό όμως δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη. Κάνοντας κάτι τέτοιο θα ε, δώσουμε μία νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για συγκεκριμένα θέματα, για θέματα ουσίας, ε, για διαδικαστικά θέματα. Εγώ θα ήθελα αυτή εξ αρχής να υπογραμμίσω την παρουσία αυτής της κοινή έκθεσης μεταξύ Ίντρε, Ίνκο και Γιούρι όπως είπαμε στη συνάντηση των συντονιστών σήμερα το πρωί, είναι σημαντικό να θυμίσουμε τη διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιτροπών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε όλα τα στοιχεία που αφορούν το διεθνές αστικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο, και το δίκαιο το που διέπει τις αγοροπολισίες θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ επιθυμώ να συμφωνήσω με τα όσα λέχθηκαν αφού πρώτα ευχαριστήσω για την έκθεση. Έχω ορισμένε παρατηρήσεις. Μιλώντας για κοινή αγορά και για να μπορέσει να λειτουργήσει η ψηφιακή αγορά πρέπει πρώτα να προστατευτούν τα δικαιώματα των δημιουργών. Η αρχή της εδαφικότητας είναι μία υπόθεση, αλλά εδώ εδαφικότητα πρέπει να βασίζεται στην έννοια του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολό της. Μόνο τότε θα έχουν και οι δημιουργοί αλλά και οι τελικοί καταναλωτές τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Βέβαια, στη βάση μιας διαφανούς νομοθεσίας. Και τα μέρη να διαθέτουν ασφάλεια δικαίου να γνωρίζουν δηλαδή ότι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά. Όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν έως τώρα στις χώρες μέλη και τις οποίες γνωρίζω θα πρέπει ωστόσο να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τις ρυθμίσεις γιατί τελείως θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ενώ τελικός μας στόχος θα πρέπει να είναι μια πλήρης εναρμόνιση, διότι αν δεν το επιτύχουμε αυτό θα συζητούμε μονάχα τις λεπτομέρειες. Για τις επιγραμμικές υπηρεσίες, online δηλαδή, νομίζω θα πρέπει να οριστούν με ακρίβεια. Όπως στο παράδειγμα των διαχειριστών ενός αυτοκινητοδρόμου που μπορεί να είναι υπεύθυνοι μοναχά για μέρος του αυτοκινητοδρόμου ανάμεσα στις πόλεις Α και Β, δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για ε, τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο. Εάν πλαστά προϊόντα κυκλοφορούν σε άλλα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, αυτά δεν μπορούν να καταστήσουν υπεύθυνο τον ε, ε, διαχειριστή ενός θυμάτου του αυτοκινητοδρόμου. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την πραγματική εφαρμογή του δικαίου και να μπορούν να αποκαλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις σαν αυτή που ανέφερα, Αυτό δεν μπορεί να βαρύνει τον διαχειριστή της επιγραμμικής υπηρεσίας αφού δεν μπορεί ο ίδιος να ε, διεξαγάγει τον έλεγχο. Γι' αυτό οι προτάσεις, οι τροπολογίες που έχουμε καταθέσει κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Αναμένω βεβαίως την περαιτέρω συζήτηση. Ε, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Άλλος κανείς, α, ο κ. Σάντερσον. Θα είμαι σύντομος. Δεν το είπαν άλλοι αυτό που θα πω. Τροπολογία δηλαδή για τα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν πρότυπα ICT τα οποία δεν είναι επαρκώς ορισμένα. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταχείριση των ευρεσιτεχνιών μέσα σε ορισμένα πρότυπα ICT, αυτό προκαλεί προβλήματα σε μικρές επιχειρήσεις και για θέματα ανοιχτής πηγής. Έχω λοιπόν ε, καταθέσει μια τροπολογία η οποία έχει το σκοπό να αρχίσει η δουλειά για να ρυθμιστεί καλύτερα το θέμα αυτό. Μάλιστα. Εσείς κύριε Λούρε, πολύ σύντομα, αφού ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, δύο πράγματα. Θα τα μεταφέρω όλα αυτά βέβαια στον κύριο Τζαμπάτσκι και το, το προσωπικό του άλλωστε παρακολούθησε τη συζήτηση, βρήκα ενδιαφέρον ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις μοιάζουν πολύ με αυτά που ακούστηκαν στη δική μου Επιτροπή Πολιτισμού. Τα θέματα είναι παρόμοια και τα επιθυμούν όλοι να καταλήξουν στα ίδια αποτελέσματα. Με ενδιαφέρει ιδίω η παρατήρηση της κυρίας Γκέριγκερ με το παράδειγμα του αυτοκινητοδρόμου. Όντω υπάρχουν αναλογίες και ίσως βέβαια προβάλλεται υπερβολικά κάπως, ε, κάποιες φορές το επιχείρημα αυτό, αλλά είναι ένα παράδειγμα το οποίο μας προσφέρει τροφή για σκέψη. Και τέλο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα βέβαια η έννοια του ασφαλού λιμένου και τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτοί που προσφέρουν περιεχόμενο, η παραγωγή περιεχόμενου δηλαδή, και η μοίρα που του επιφυλάσσεται. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, έχουμε τώρα ολοκληρώσει το υπαριθμό 13. Ακολουθεί το 14. Ανταλλαγή απόψεων για περιόδους περιορισμού για τροχαία ατυχήματα. Εδώ είμαι εγώ ο ίδιος εισηγητής, αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι μία παρεμφερής έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Αυτή ξεκίνησε το 2006 από την ε, Επιτροπή Νομικών Θέσεων και αφορούσε τι ακρατικές διαφορές που κατέληγαν σε θανατηφόρα ατυχήματα. Η συγκίτρια ήταν η κυρία Νταϊάννα Βόλις. Μετά κολούθησε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο του 2007. Η έκθεση αυτή ζήτησε από την Επιτροπή και παραθέτω να προβεί σε μία έρευνα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της περίοδου ρυθμού της εσωτερικής αγοράς και ιδιαίτερα ως, σε ό,τι αφορά τους πολίτες που ε, καλύπτονται από την συνθήκη. Η Επιτροπή θα έπρεπε να καθορίσει ποσοτικά τις περιπτώσεις τραυματισμών και να αξιολογήσει δυσκολίες ε, τρίτων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποιος σαν αποτέλεσμα ε, αλλαγών στην περίοδο και στις δυνατότητες που κυμαίνονται μεταξύ περιορισμένης εναρμόνισης μέχρι ε, της ε, περίπτωσης όπου υπάρχει σύγκρουση δικαίου. Τέλος, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων. Η Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό ξεκινώντας μία μελέτη σχετικά με την αποδημίωση των θυμάτων που είχαν εμπλακεί σε θανατηφόρα ατυχήματα. Μία σύγκριση των πρακτικών, ανάλυση των προβλημάτων και των επιλογών σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, μιλάμε πάντοτε για την περίοδο παραγραφής, για την προθεσμία παραγραφής. Σε αυτή τη μελέτη αναφέρθηκε πρώτον ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά το καθεστώς παραγραφής και εν ώψη αυτού υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος εκτροπών. Υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών που κινούνται από μια ε, εθνική προσέγγιση μέχρι την εισαγωγή, μέχρι την δημιουργία ενός ανευρωπαϊκού δικαστηρίου που θα ακολουθήσει τους κανόνες, που τους υπάρχοντες κανόνες για την περίοδο παραγραφής. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει οργανώσει δύο διαβουλεύσεις, μία το 2009 και μία άλλη το 2012 με σκοπό να εντοπιστούν τα εμπόδια ή τα θύματα διακρατικών ατυχημάτων στις περιπτώσεις εκείνες που προσπαθούν, που επιδιώκουν να λάβουν μία αποζημίωση για ζημίες που έχουν υποστεί. Το 2012 η τα κατά διάρκεια των διαβουλεύσεων οι εμπλεκόμενοι εκλήθησαν να εξετάσουν διάφορους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Πρώτον, το ε, να, να υπάρχει καλύτερη ε, πληροφόρηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεύτερη επιλογή, να βελτιωθεί να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για αντικείμενα που έγιναν στο εξωτερικό και αυτό να θεωρηθεί υποχρεωτικό. Τρίτη επιλογή, να, υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες ότι αφορά την περίοδο παραγραφής. Τέταρτη, δυνατότητα εισαγωγή νέων κανόνων εναρμόνισης της περίοδου παραγραφής σε περιπτώσεις διακρατικών τροχαίων. Η Επιτροπή παρόλα αυτά Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση σε αυτό το τομέα. Ο στόχος ε, της ε, της ε, έκθεσης είναι να τεθεί και πάλι το θέμα επιτάπητος και να υπάρξει μια σύσταση στην οποία, η οποία πείσει την Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος. Στην όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η παραγραφής παίζουν καθοριστικό ρόλο και ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το 2011 η πρόσβαση σε εκθέσεις της δικαιοσύνης από πλευράς της, ε, ε, ε, της αρχής ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέληξε στο ότι αυτά είναι αναγκαία για να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου αυτές οι διαμάχες. Αυτά τα συμφέροντα θα πρέπει να εξισορροπούνται με το βασικό, με το θεμελιώδες δικαίωμα να αποζημίωσης από τη στιγμή που με ένα σύντομο διάστημα παραγραφής θα μπορούσε να παρακολύσει την απονομή δικαιοσύνης. Με βάση αυτό Υπάρχουν δύο σημαντικέ παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, οι περίοδοι παραγραφής ποικίλουν μεταξύ των χωρών μελών, ενώ τα νομικά καθεστώτα στην υπηρετική Ευρώπη αναφέρονται σε περιόδους παραγραφής, prescription period, δηλαδή μετά την εκνοή των οποίων μπορεί να ε, υποβληθεί ένα αίτημα σε χώρες του εθνικού δικαίου υπάρχουν περίοδοι παραγραφής που αναφέρονται στον χρόνο μετά τον οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα προβολής ε, απαιτήσεων. Υπάρχουν διαφορές ε, και στις περιόδους παραγραφής σε ό,τι αφορά την αρχή της περίοδου στην περίπτωση αναπήρων και ανηλίκων. και αυτό ως, ως, τη δυνατότητα διακοπής της περίοδου παραγραφής. Δεύτερον, στα διακρατικά τροχέα τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή αιτήματος καθορίζονται από τους νόμους του κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα το τροχαίο Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού, η εθνικοί νόμοι για την περίοδους παραγραφής είναι πολύπλοκοι και τα θύματα πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τους κανόνες της χώρας μέλου, μέλους στην ε, οποία ταξιδεύουν. Αυτό σε συνδυασμό με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των νόμων περί παραγραφής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις για τα θύματα και να δημιουργήσουν πάρα πολλά εμπόδια σε ό,τι αφορά το δικαίωμα σε αποκατάσταση και σε έγκαιρη ε, και εύλογη ρύθμιση ε, του, ε, της δαφάνης. Ε, επικοινωνήσαμε με την κυρία Τζέννη Παπαδά και ζητήσαμε να κάνει μια μελέτη σχετικά με την προστιθέμενη αξία της νομοθετικής πράξη στον τομέα των περιόδων παραγραφής για διακρατικά τροχέα. Η τελική μελέτη θα υποβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου και θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές ε, ακροάσεις Αυτή η ακρόαση προβλέπεται να γίνει το πρώτο εξάμεινο του 2016 και θα πάρουν μέρος διάφοροι σχετικοί φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτά είχα να σας πω και ελπίζω να ακολουθήσει μία ενδιαφέρουσα συζήτηση και συνεργασία. Παρακαλώ. Το λόγο έχετε εσείς τώρα σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια σύσταση ή αν έχετε να κάνετε κάποια ένσταση. Mr. Le Ο κύριος Λεμπρετών. Προσωπικά πιστεύω ότι το πρόβλημα των αποζημιώσεων σε οδικά και τροχιά αντικείμενα, παρόλο που έχει διασυνοριακά χαρακτηριστικά, ε, είναι αρμοδιότητα κρατών μελών. Μεταξύ των λύσεων που έχετε προβάλει, προτιμώ μία ξεκάθαρα, μακράν. Είπατε ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές λύσεις, εγώ προσωπικά βλέπω μόνο δύο. Μπορούμε να επιλέξουμε δύο λύσεις ή θα βελτιώσουμε την πληροφόρηση με τρόπους εφαρμογής που θα επινοήσουμε στη συνέχεια ή θα εναρμονίσουμε τους νομικούς κανόνες για την περίοδο παραγραφής, το χρονικό όριο. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κλείνουμε προς την πρώτη λύση, δηλαδή να βελτιώσουμε την πληροφόρηση, αυτό θα φτάσει και θα περισσέψει για να, ε, και θα μπορέσουμε έτσι να επιλύσουμε τα προβλήματα. Η κυρία Ντελβό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν κατάλαβα καλά, εσείς ως εισηγητής συντάσσετε αυτή την έκθεση για να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει το βήμα της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη διαπιστώσει ότι είναι επίγον βεβαίως, ότι ε, πρέπει να δράσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι βεβαίως δεν επιθυμούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη την πλήρη εναρμόνιση. Όμως, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίποτα θα μας εμποδίζει να καταλήξουμε σε συστάσεις και να πούμε ότι, για παράδειγμα, ε, το ελάχιστο χρονικό περιθώριο, η μίνιμουμ προθεσμία θα είναι αυτή ή ότι θα υπάρχει, μας ένας ελάχιστος συντονισμός καλές οι πληροφορίες, αλλά πολύ συχνά ενδιαφέρεται ο κόσμος να ε, συλλέξει τις πληροφορίες μόνο όταν είναι ήδη πολύ αργά. Ε, είναι δύσκολο να είναι κανείς καλά ενημερωμένος εκ των προτέρων. Θεωρώ λοιπόν ότι ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ακριβώς να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Διαπιστώνοντας λοιπόν ότι οι πολίτες μετακινούνται όλο και περισσότερο και ε, περνούν από τη μία μεριά των ε, εθνικών συνόρων στην άλλη όλο και περισσότερο, ε, τέτοιου είδους βοήθεια είναι εξαιρετικά χρήσιμη στους χρήστες των ε, οδών, του οδικού δικτύου των χωρών. Χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ και βεβαίως ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας με, πάνω σε αυτό το φάκελο. Δεν βλέπω να ζητά κανείς κάποιος άλλος τον... Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλος τον λόγο. Μπορούμε να θεωρήσουμε λήξα σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και να προχωρήσουμε στο σημείο 18, ανταλλαγή απόψεων ε, για την αντιπροσωπεία που μετέβει στο Κίεβο στην Ουκρανία για την αντιπροσωπεία στο Κίεβο. Ίσως εγώ μπορώ να ενημερώσω για αυτή την αποστολή, ε, να πω στα παρόντα μέλη ότι τέσσερις ήταν αυτοί που αποτελούν μέρος της αποστολής, κυρία Χαουτάλα, κυρία Μπερζεγόν, κύριο Σουτσπάτσκι και ο υποφαινόμενος. στόχος της αντιπροσωπείας ήταν με βάση τις δικές μας αρμοδιότητες για δικαστική συνεργασία σε θέματα ε, αστικού δικαίου, ε, πολιτικής δικονομίας και με βάση τις λοιπές αρμοδιότητες που έχουμε στον τομέα αυτό, ε, πήγαμε στο Κίεβο, στην Ουκρανία, για να δούμε τις διαδικασίες τις διαδικασίες κύρωσης της συμφωνίας με, την Ουκρανία, η οποία συμφωνία ε, πλησιάζει η λήξη της και η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώθηκε στην πιο επίκαιρη χρονική στιγμή, στην πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία, γιατί ε, διαρθρώνεται και μεταρρυθμίζεται ρίζοσπαστικά το δικαστικό ε, σύστημα στην Ουκρανία και αυτή την προσπάθεια την επικουρεί μία συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταρρύθμιση, ε, την τομεακή, την δικαστική στην Ουκρανία. Είναι η EU η οποία είναι παρούσα από τον Ιούλιο του 2014 στη χώρα αυτή. Η μεταρρύθμιση είναι ρίζοσπαστική πραγματικά και είχαμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε με τα μέλη του, του, της Φερκόφνα Ράντα του Ουκρανικού Κοινοβουλίου με μέλη ε, και του συνασπισμού που βρίσκεται στην κυβέρνηση αλλά και με μέλη της αντιπολίτευσης. Επομένως, ακούσαμε όλες τις ε, γνώμες και τις απόψεις ε, για αυτή τη μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα, η αποστολή έλαβε χώρα με παράλληλη ε, αποστολή από την Επιτροπή Ίντα η οποία ασχολείται με τις ε, σχέσεις ε, με το εξωτερικό εμπόριο. Ταυτόχρονη λοιπόν διοργάνωση αυτών των αποστολών είχε νόημα αυτή η κοινή, η αποκοινού διοργάνωση, διότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ουκρανία είναι καθοριστική για τους ενδυνάμει επενδυτές για να επενδύσουν στην Ουκρανία. Έχει δηλωθεί ότι μόνο μετά την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης οι επενδυτές θα έχουν εμπιστοσύνη ότι μπορούν να επενδύσουν στο ουκρανικό έδαφος. Και πέρα από τις συναντήσεις ε, στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, στη Βερκόφνα Ράντα. Συναντηθήκαμε επίσης με τον πρόεδρο και τους συναδέλφους μας από το ανώτατο Ουκρανικό Δικαστήριο. Είχαμε μία ε, συνάντηση μίας ώρας με τον πρόεδρο Ποροσέγκο και Είδαμε και την ε, άρτη συσταθήσα και ιδρυθήσα υπηρεσία πολέμησης της διαφθοράς. Ήταν πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμα της αντιπροσωπείας μας. Ε, ούτε καν προλάβαμε να φάμε μεσημεριανό φαγητό τις περισσότερες φορές. Είχαμε, γιατί είχαν παρευληθεί πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις επί τόπου. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να βοηθήσω την κυρία Χαουτάλα, να εκφράσω τη στήριξή μου στην άποψή της η οποία ε, λέει ότι αφού η αποστολή αυτή ήταν τόσο σημαντική, τότε η δική μας Επιτροπή να εξετάσει και παρεμφερείς αποστολές και αντιπροσωπείς σε σχετικές συνδεδεμένες χώρες. Επομένως συμφωνώ με αυτή την πρόταση και ε, σας ευχαριστώ Γεωργία. Αυτά είχα να σας πω από την πλευρά μου. Κοιτάζω λίγο και το Χάραλντ ε, να δω αν έχω ξεχάσει κάτι σημαντικό που δεν είπα στα μέλη. Τι λέτε. Όχι. Καλώς. Ε, τα μέλη της Επιτροπής μας έχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, ε, είναι η ώρα να πάρετε το λόγο γιατί από την τετραμελή αντιπροσωπεία εγώ είμαι ο μόνος που είμαι παρόν αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας κατατοπίσω. Ο κύριος Κέστερ. Έχω μια ερώτηση, ωστόσο κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σφόβοντα, περιγράψατε διάφορα θέματα που συζητήθηκαν σε διάφορες συσκέψεις. Ποια είναι ωστόσο η τελική σας άποψη. Θεωρείτε ότι η Ουκρανία προχωρεί προς την υλοποίηση ενός αξιόπιστου ε, κράτους δικαίου και δημοκρατικών θεσμών, διότι διαβάζω στον τύπο ότι υπάρχουν και ισχυρές εθνικιστικές και εν μέρη και φασιστικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ε, ποια είναι τελικά η άποψή δηλαδή η τελική σας άποψη, πού βρίσκεται η Ουκρανία, ο πρόεδρος Βόμποντα. Γνωρίζετε ότι αυτές που αποκαλείται φασιστικές δυνάμεις απέτυχαν στις ε, πιο πρόσφατες εκλογές. Άρα η πολιτική τους επιρροή είναι ελάχιστη. Και οφείλω να πω κιόλα ότι η νομοθετική πλευρά αυτή της δικανική μεταρρύθμιση είναι αρκετά θαραλέα. Και εάν υλοποιηθεί ορθά, θα σημάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Στην κατεύθυνση της θέσπισης ενός πραγματικού κράτους δικαίου. Δηλαδή, η Ουκρανία ολοκληρώνει τώρα την νομοθετική διαδικασία και βέβαια τώρα θα έλθει η φάση της υλοποίησης. που και αυτή φαίνεται ότι αποτελεί πρόκληση και το λέω βέβαια ε, και με τριοπαθός. Μάλιστα, και ορίστε κύριε Κρέστερ. Μία ακόμη ερώτηση. Ένα σημαντικό θέμα στην Ουκρανία είναι και ο ρόλος της Ανατολικής Ουκρανίας. Εκεί προσπαθούν να φτιάξουν ένα μάλλον ομοσπονδιακό σύστημα όπου οι περιφέρειες ε, θα έχουν μεγαλύτερη αυτονομία. Αυτό το στοιχείο έπαιξε στις ε, συζητήσεις σας κάποιο ρόλο. Ο πρόεδρος Φόμποντα. συζητήθηκε μεν το θέμα αυτό, αλλά όχι σε βάθος. Αναφέρθηκε μόνο όταν ομιλούσα για επενδύσεις στην Ουκρανία. Ακόμη δηλαδή και το γεγονός ότι το ανατολικό μέρος της χώρας είναι αποσταθεροποιημένο σε ένα βαθμό, ότι το γεγονός αυτό δεν θα πεθάρινε κατά βάση πιθανούς επενδυτές από την υλοποίηση επενδύσεων και ότι το βασικό πρόβλημα είναι η κατάσταση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Δεν συζητήσαμε όμως ευρέως το πρόβλημα της Ανατολικής Ουκρανίας. Δεν βλέπω άλλους ερωτώντες. 19. Είμαι πάλι συζητής για το 19 και για να κάνω τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα θα αρχίσω να σας μιλώ τσεχικά. Ε, ε, Ευχαριστώ λοιπόν που με επιτρέπετε να συνεχίσω. Ορισμένοι εξημών έχετε ήδη συμμετάσχει σε συζητήσεις για το θέμα της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας Επιτροπή καλείται να συντάξει μια γνωμοδότηση, αν και η αρμόδια επιτουσίας Επιτροπή είναι η Επιτροπή των Συνταγματικών Θεμάτων. Είναι βεβαίως σημαντικό αυτό όσον αφορά τη θετική εικόνα προς τα έξω των ευρωπαϊκών θεσμών και για να συμβάλλουμε στη δημιουργία αυτής της ε, διαφάνειας είναι σημαντικό να εργαστούμε για τη διεύρυνση του θέματος. Η διαφάνεια για μένα δεν είναι εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα. Τα βήματα που πρέπει να κάνουν τα διάφορα θεσμικά όργανα νομίζω προσεκτικίνες τώρα νομίζω ότι βαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Βέβαια χρειάζονται ε, μεγαλύτερη επεξεργασία. Πρέπει να δούμε τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται στις συνθήκες. Στη συζήτηση συζητήθηκε το θέμα, ναι, το άρθρο μάλλον 15, της, ε, το άρθρο 15 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί λέει ότι στόχος είναι η σωστή, η ορθή διαχείριση των θεμάτων με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ε, οι θεσμοί και τα άλλα όργανα πρέπει να είναι ανοιχτά σε αυτή την προσπάθεια. Στην παράγραφο του 3, του άρθρο 15, λέει ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης και κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί η κατοικεί σε μια χώρα μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στους θεσμούς και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέει, η, αυτά το οικείο αυτό άρθρο της ε, συνθήκης. Και αυτά έχουν συζητηθεί και σε ακροάσεις και σε μελέτες. Και μάλιστα και σε ακρόαση όπου είχαμε οργανώσει εμείς οι ίδιοι και όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την κατάσταση όπως αυτή είναι σήμερα και μάλιστα υπάρχει και περιθώριο για να συνταχθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας. Χρειάζεται να εγγύψουμε στη διαφάνεια και σε ευρύτερο επίπεδο αλλά και ιδίως στα θέματα εκείνα που απλήττουν των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Για παράδειγμα, έκδοση εγγράφων έτσι ώστε ε, η γνωμοδότηση να συνταχθεί με έναν υφάλιο τρόπο. Αναμένω δυσικές προτάσεις και είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας για την τελική μορφή της ε, εκθέσεως και ελπίζω να είναι και θετικό το αποτέλεσμα. Σε αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα, το, το σχέδιο της νομοδοτήσεως θα πρέπει να υποβληθεί στις 12 ενδεκάτου. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 19 ενδεκάτου ψηφοφορία στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Δεκέμβριο στο Στρασβούργο. Αυτά όλα είναι όλα από την πλευρά μου. Βέβαια ε, είναι κρίμα που δεν είναι παρούσα η κυρία Χάουταλα που ε, σίγουρα ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη συζήτηση και ασφαλώς έχει μπορά να ε, συμβάλλει. Πάντως αναμένω τη συζήτηση μαζί σας και τη σχόλιά σας. Αυτά λοιπόν στα τσεχικά και τώρα συνεχίζω στα αγγλικά και περιμένω βεβαίως να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ε, well, I do not... Δεν βλέπω κανένας να ζητεί το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι λίγη εδώ η ανταλλαγή απόψεων, αλλά ανταλλαγή απόψεων εγώ την ερμηνεύω αυτήν ως πλήρη συνένεση στα όσα σας είπα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήλθατε και συναντηθήκαμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε στις